Χριστίνα. Και καλωσορίσατε σε αυτό το διάλογο των πολιτών. Και τώρα πραγματικά έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε στον Επίτροπο Τίμπορν Νάβατσιτς. Να τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται μαζί μας σήμερα και για τον διάλογο αυτό ή το θέμα της, τέχνο, δημοκρατίας, τη δημοκρατία και εγώ. Να σας υπενθυμίσω ότι είστε υπεύθυνοι σε θέματα εκπαίδευσης, παιδείας, νεολαίας, αθλητισμού. Είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την νεολαία και γι' αυτό Θέλουμε κατεξοχήν με εσά να μιλήσουμε. Τα επόμενα 90 λεπτά θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον Επίτροπο, ο οποίο θέλει να ακούσει τι απόψει σα. Πώ ε, Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο στη ζωή σας. Οι ευρωεκλογέ, οι ευερχόμενες έχουν σημασία για σας. Μπορεί να θέλετε να μας μιλήσετε για τις ελπίδες σας, για τις ανησυχίε σας, τους φόβους σας για το μέλλον. Και είσαστε νέοι, είσαστε από τόσες πολλές χώρες, έχετε τόσο διαφορετικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε live στο ημικύκλιο εδώ. Είμαστε ένα μοντέλο δημοκρατίας και θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις σας. Φυσικά, να πάρετε όλοι το λόγο, όχι μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα και φυσικά όσοι έχουν ήδη πάρει το λόγο να ξαναπάρουν το λόγο αν το επιθυμούν. Στα αγγλικά μπορείτε να πάρετε το λόγο ή σε οποιαδήποτε από τις 22 άλλες επίσημες γλώσσες είναι αυτή η ομορφιά της Ευρώπης. Να ευχαριστήσω τη στρατιά των διερμηνέων που είναι μαζί μας σήμερα. Τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Just a couple of words about my πω δύο λόγια για το δικό μου ρόλο συντονιστή. Θα ήθελα λοιπόν να εξασφαλίσω ότι θα πάει καλά η ανταλλαγή αυτή απόψεων. Όταν θέλετε λοιπόν να μιλήσετε, να σηκώνετε το χέρι σα και θα σας δίνουμε το λόγο. Έχετε και το κόκκινο κουμπί για να ανοίξετε το μικρόφωνο. Να μας πείτε το όνομά σα, να μα πείτε από πού είσαστε. Και τέλος, να είσαστε σχετικά σύντομοι σε αυτά που λέτε. Όχι μόνο μία πρόταση, θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε, αλλά θέλουμε να πάρουν και όλοι το λόγο, όσοι το επιθυμούν. Και τέλος, να ευχαριστήσω όσους συμμετέχουν online στην ιστοσελίδα μας ή μέσω του Twitter. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν τώρα δύο hashtags σήμερα. Youth Week Χρησιμοποιήστε το όσο θέλετε λοιπόν. Έχουμε και το hashtag EU Dialogue. Καλά ορίζουμε τα σχόλιά σας. Λοιπόν, έχουμε και το τηλέφωνο εδώ, το έχω πρόσφατα, το έχω κοντά μου και μπορώ να τσεκάρω. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πείτε, να σας ε, ε, παρουσιάσω τον κύριο Μέιπελ από την Νάπολη ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη για να συναντηθεί και με άλλους νέους. Ο κύριος Ρούσο ε, και μαζί ε, μα εξερεύνησαν το ευρωπαϊκό τοπίο. και Ας δούμε αυτό το βίντεο λοιπόν. But firstly, it was a unique opportunity. The opportunity to explore other cities, to meet other people on the road, and magically transform strangers into new friends. But we surely asked,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 Να ξεκινήσουμε για να ακούσουμε και πιο πολλά για αυτή την ε, πολύ όμορφη πρωτοβουλία Discovery You. Αλλά πρώτα να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Ναβατσίτς για να ανοίξει και επίσημα την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Good morning and thank you very much. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό ε, γεγονό. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για του νέου, αλλά και για του πολιτικού ευθύνοντε, για όλα τα άτομα εκείνα που καθορίζουν το μέλλον μα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή η εβδομάδα τη νεολαίας, γιατί μένουν τέσσερι εβδομάδε μέχρι τι ευρωεκλογέ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν μπορεί κανείς λοιπόν να εκφράσει την άποψή του για το μέλλον, όταν ψηφίσει για να διαμορφώσει πραγματικά το μέλλον. Πριν από πέντε χρόνια, όταν ξεκίνησα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλειδονίζονταν από οικονομική κρίση και το επίπεδο της ανεργίας στους νέους σε κάποιες χώρες ήταν πάνω από 50%. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση αυτή. Κάποιοι προβλέπουν νέους κλειδονισμούς για το φθινόπωρο αλλά προς το παρόν πρέπει να σας πούμε ότι μάλλον βγαίνουμε από την πιο σημαντική φάση της οικονομικής αυτής κρίσης. Θα πρέπει να συζητήσουμε όμως τις μεραντικές πτυχές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για σας προκειμένου να αισθανθείτε ασφαλείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπουμε πολλές συζητήσεις και πολλές συγκρούσεις σε πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κρατη θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Να τα συζητήσουμε για να θέλουμε ένα μήνυμα στους πολιτικούς και στους μελλοντικούς πολιτικούς για τις δικές σας προοπτικές. Αν μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τις δικές σας απόψεις, το δικό σας feedback για το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε από κοινού να κάνουμε κάτι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Καλώς ορίσατε και πραγματικά χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Ελπίζω να είναι πολύ α, επικοδομητική η σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, Commissioner. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε μέσα στο διάλογο. Ποιος θέλει να σπάσει τον πάγο. Εσείς σηκώσατε πρώτο στο χέρι, εσείς έχετε πρώτο στο λόγο. Ευχαριστώ, αλλά θέλω να τα πω μαλτέζικα. Λυπάμαι, λυπάμαι, χίλια συγγνώμη από τις πολύ λίγες γλώσσε που δεν μπορούμε να καλύψουμε σήμερα. Καλά τότε να μην επαναλάβω. Έχουμε μαλτέζικα. Έχουμε μαλτέζικα, με συγχωρείτε. Ε, λάθος πληροφορία, μπορείτε να μιλήσετε μαλτέζικα. Αυτό που θέλω να πω είναι απλό. Είπατε, Επίτροπε, ότι θέλετε δουλειά, απασχόληση για τους νέους. Ερώτηση. Γιατί δεν βρίσκουμε όμως νέους μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των πολιτικών εθνόντων. Και επίσης γιατί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο Έχουμε ε, σταζιέρ που δεν έχουν αρκετά για να πληρώσουν τον νίκη τους, που δεν, ε, πληρών, δεν παίρνουν αρκετά. Πώς δίνει το παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς εσείς δίνετε το παράδειγμα χωρίς να επιτρέπετε στους νέους ε, να ε, συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. yes, ναι, για τη συμμετοχή των νέων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, είναι πολύ ευρή ερώτηση ως πρώτη. Θα μπορούσα να σας παρουσιάσω ένα πολύ συνολικό πλαίσιο για την ε, συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη. Όμως οι νέοι πρέπει να ψηφιστούν. Οι ψηφοφόροι αποφασίζουν αν θα έχουμε νέο στην πολιτική. Πρέπει να σας ψηφίσουν ε, οι ψηφοφόροι για να αποφασίσουν αν θα είστε βουλευτή στη Μάλτα ή εδώ σε αυτό το μεκύκλιο του Στρασβούρκου των Βρυξελών. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας με τους νέους. Κοινωνικό διάλογο θέλουμε με τα θεσμικά όργανα, την τα κλασική διαδικασία διαλόγου αλλά τώρα θέλουμε να καταφέρουμε να συγκινήσουμε τους νέους που δεν είναι μέλη καν ενώσεων νέων, που δεν εκπροσωπούνται από ενώσεις νέων. Γιατί αυτούς κάπου χάνουμε στο δρόμο. Είναι απομονωμένοι, ε, μονάδες, γίνονται μονήρις. Αυτούς πρέπει να εντοπίσουμε λοιπόν στην όλη προσπάθεια, να τους καλέσουμε στο κέντρο της κοινωνίας. Διότι Εάν με τα δικαιώματά τους πάνε σε εκλογικό κέντρο στο τέλος Μαΐου για να ψηφίσουν, ποιοι θέλουν να τους εκπροσωπήσουν ή να είναι οι υποψήφοι, θα πρέπει οι φωνές τους να ακουστούν και σε πιο θεσμικό επίπεδο. Κατά τα άλλα έχουμε και πολλά προγράμματα. Το πιο, το πιο γνωστό είναι το πρόγραμμα μαθητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι έξι μήνες ε, στάζ αυτό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ καλοπληρωμένο. Μπορεί κανείς να έρθει εδώ, μπορεί να εξοικειωθεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και μετά ίσως να βρει και δουλειά. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, να σας προσφέρουμε ευκαιρίες εσάς τους ενεργούς νέους για να μπορείτε να συμμετέχετε στι ευρωπαϊκέ διαδικασίε ή τέλο πάντων σε όσα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σας ευχαριστώ. Έχουμε και εδώ μια ερώτηση. Είμαι η Ντάρο και, θα... και με τη θα μιλήσω αγγλικά για να κάνουμε πιο γρήγορα. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι στην πολιτική, όχι γιατί δεν συμμετέχουν στο διάλογο. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπατε και προηγουμένω, το τι θα γίνει με τους νέους και αν πάνε να ψηφίσουν. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τους πολιτικούς. Δεν πρέπει να συμμετέχουν στον διάλογο και σε ένα επίπεδο λήψης αποφάσεων. Μα πάντα δουλεύουμε με νέους. Εγώ όταν ήμουν υπουργό μεταξύ του 2007 και του 2014 είχα μεταξύ των συνεργατών μου δύο τρίτα κάτω των 35. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί να προσφέρουν τις ευκαιρίες και να καλλιεργήσουν τη σχέση με τους νέους. Για μένα δεν είναι καν πολιτικό ζήτημα, είναι ευαισθησία. Ευαισθησία προς τους νέους. αλλά δεν υπάρχει κάποια γενικευμένη λύση. Μπορούμε να βρούμε μια ποσόστοση για τους νέους, αλλά δεν θα ήταν λύση, θα ήταν διοικητικό το μέτρο. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους πολιτικούς ότι οι νέοι δεν είναι απώλεια, είναι επένδυση για το μέλλον. Αλλά διαρκώ νομίζω υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό. Αν ρωτήσετε του βουλευτέ σα, θα ανακαλύψω ότι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο περισσότεροι μεταξύ των συνεργατών, των βοηθών, των ειδικών περιπολιτική. είναι νέοι. Εγώ βρίσκω ότι υπάρχει διαφορά. Μπορεί να μην πηγαίνει αρκετά γρήγορα, αλλά υπάρχει εξέλιξη. Θέλει και λίγο απομονή. Βεβαίω πρέπει να πείσουμε τους εμπειρότερους πολιτικούς να προσλάβουν νέου. Καλημέρα. Επίτροπε. Είμαι ο Ρικάρντο από την Ιταλία και θα μιλήσω αγγλικά. Μ' αρέσει που ο καθένα μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά μ' αρέσει να μπορώ να μιλήσω και τα αγγλικά, γιατί θέλουμε να είμαστε ενωμένοι στην ποικιλομορφία. Και είναι ένα τρόπο να ενωθούμε γλωσσικά αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτή η συγκέντρωση, αλλά υπάρχει κάτι που με ενοχλεί η επανάληψη του όρου ε, νέοι. Ξέρω την εβδομάδα των νέων, αλλά όπως και με το φίλο, ε, νομίζω ότι είμαι απλώς ένας πολίτης που ε, τυχάνει να είμαι νέος. Δεν μπορώ να ταυτιστώ λοιπόν με όλες τις ηλικίε, ξέρω εγώ αυτούς που είναι 135 ότι υποτίθεται ότι θεωρείται νέο. Η κοινωνία των πολιτών μαζί με τους πολιτικούς θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο στην αξιοκρατία παρά στην ηλικία ή το ποσό της ε, πείρας. Ποιοι είναι λοιπόν οι διάβλοι από τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε τις ικανότητές μας. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο, παρά η ηλικία από την οποία μπορεί κανείς να αρχίσει να έχει πρόσβαση στην πολιτική και μετά. Η ερώτησή σας να οδηγήσει στο διαρκέ πρόβλημα τη πολιτική για τους νέου. Δηλαδή, εάν η πολιτική για τους νέου είναι ξεχωριστός ε, πολιτικός χώρο ή πρέπει να είναι οριζόντια διάσταση. Η διάσταση των νέων να υπάρχει σε όλες τις πολιτικές. Νομίζω και τα δύο είναι σημαντικά. Διότι από τη μία αυτό που κάνω είναι να συμπεριλάβω τις πτυχές για τους νέου σε όλα τα κομμάτια όλων των πολιτικών διότι όπω σωστά λέτε είναι απλώ ομάδα ηλικιακή οι νέοι. Από την άλλη όμω υπάρχουν ειδικέ ανάγκες που εκπροσωπούνται καλύτερα Εάν δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή τη ηλικία ομάδα, λόγω χάρη, πρώτη δουλειά, πρώτη οικογένεια, πρώτο σπίτι, Πρέπει λοιπόν να δούμε τις ανάγκες της ηλικιακή αυτής ομάδας για να εντοπίσουμε τι χρειάζεται. Ε, είναι Ευρωπαίοι πολίτες οι νέοι, δεν είναι απλώς νέοι. Έχουμε και άλλε όμω εκδηλώσει. Εκεί επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ιδιότητα του πολίτη. Και συμπεριλαμβάνουμε νέου. Συμπεριλαμβάνουμε τη διάσταση των νέων ε, για το, στο πλαίσιο τη κοινωνία των πολιτών. Εδώ μας ενδιαφέρουν οι δικές σας ανάγκες και θέλουμε να συζητήσουμε τα δικά σας ιδιαίτερα προβλήματα και να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Εσείς είστε το μέλλον σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια θα έχετε θέση λήψης αποφάσεων. Εσείς θα ηγείστε στην ευρωπαϊκή οικονομία, πολιτική, πολιτικό, πολιτιστικό βίο, παντού. Ε, θα πρέπει να μιλάτε μεταξύ σας, να συνεννοείστε και να μας ενημερώνετε ποιες είναι οι απόψεις σας ε, τι θέλετε εσείς ως Ευρωπαίοι για το μέλλον για να προετοιμαστεί το μέλλον ήδη με τις σημερινές μας αποφάσεις πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ μια ερώτηση από πίσω τώρα. Από τις πίσω σειρές. Εσείς κυρία μου, εκεί πίσω. Ναι, ναι, εσείς. Όχι, όχι, ναι, ναι. Η Λίζα είμαι από την Αυστρία. Και εγώ έχω έρθει σήμερα με τους συναδέλφους μου Έχουμε μια ε, οργάνωση νεολαία. Οι νέοι λοιπόν ενδιαφέρονται πολύ για την πολιτική, θέλουν να παρακολουθήσουν την πολιτική, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ε, τολμούν να ψηφίσουν. Α, συγγνώμη, δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν. Δεν, τους, ε, δεν έχουν δικαίωμα να παρουσιαστούν στις εκλογές. Είναι πολύ μεγάλο θέμα λοιπόν αυτό, ότι δεν ακούγεται η φωνή των νέων γιατί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.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 και το θέμα των προσφύγων που επηρεάζονται από την ε, νομοθεσία ε, αλλά δεν ε, μπορούν να ψηφίσουν οι πρόσφυγες να καθορίσουν την πολιτική, αλλά τους ενδιαφέρει η πολιτική. Είναι πολλοί νέοι που τους ενδιαφέρει η πολιτική και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλλά το δικαίωμα του, της ψήφου συνδέεται πάντα με το θέμα της ηθαγένειας και της ποιότητας. Μόνο το σοβιετικό αμα, Σύνταγμα το 1918 δεν συνέδεσε το δικαίωμα ψήφου με την υπηκότητα, με την ηθαγένεια, αλλά μόνο με την ταυτότητα της τάξης μπορούσε να ψηφίσει όποιος ήθελε και όποιος ήταν σοβιτικός. Αλλά συνήθως ε, συνδέεται με το θέμα της ηθαγένειας. Ένας ε, πρόσφυγας μετανάστης, ο οποίος καταφτάνει σε μια χώρα και έχει ηθαγένεια, μπορεί να ψηφίσει. Αν δεν έχει ηθαγένεια, δεν μπορεί να ψηφίσει πολύ, φοβάμαι. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε λοιπόν αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κάθε μελη πρέπει να αποφασίσουν ποιο έχει δικαίωμα ψήφου και ποιο όχι. Και θα ζητήσω από τους τεχνικούς μας να τσεκάρουν λίγο τα ακουστικά μας, γιατί δεν ακούσαμε την ερμηνεία. Στην uh, θέση 61 να ακούσουμε. Okay, so I'll try in English. So when I go to school in the morning... Όταν πηγαίνω στο σχολείο το πρωί είναι 8 το πρωί και επιστρέφω στις 6 το απόγευμα. Σε 10 ώρες λοιπόν χρησιμοποιώ την Ευρώπη και ξέρω ότι συμμετείχα στην Ευρώπη. Αν δεν είχα συμμετέχει σε προγράμματα όπως το Erasmus Plus και αν δεν υπήρχαν τέτοια προγράμματα, αναρωτιέμαι τι πλεονεκτήματα θα είχα από την Ευρώπη. Δεν θα τα ήξερα. Για 10 ώρες λοιπόν θα είχα αξιοποιήσει την Ευρώπη και δεν θα το ήξερα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι πάντα εκεί και έχει γίνει κάπως ε, φυσιολογικό και φυσικό να υπάρχουν τα πλενεκτήματα που έχουμε από την Ευρώπη. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι όλα αυτά τα πλεονεκτήματα θα υπήρχαν και χωρίς την Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Ο κόσμος θεωρεί ότι «Ε, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Μια χαρά είμαστε. Αλλά έχουμε τα πλεονεκτήματα. Και θα συνεχίσουμε να τα έχουμε. Αυτό δεν εκεί όμως. Εγώ από πλευρά μα να σα πω ότι είμαστε 90 μαθητέ στη χρονιά μου και νομίζω ότι 6 πραγματικά ξέρουν τι κάνει η Ευρώπη. Την πρώτη φορά που άκουσα για την Ευρώπη ήμουν 8 χρονιών. Κάναμε κάποια μαθήματα και μετά τίποτα. Ούτε ξανακούσαμε το θέμα της Ευρώπης. Εγώ συμμετείχα στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εβδομάδα Νεολαία και ενημερώθηκα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υπόλοιποι όμω 84 τη χρονιά μου δεν ξέρουν τίποτα για την Ευρώπη. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Πώ μπορούμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Από πού είσαστε, για πείτε μου. Από τη Γερμανία, από τη Γερμανία, ναι, ναι. ναι. I totally agree with you and I... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Μακάρι να την ήξερα, το πρόβλημα θα ήταν λυμένο αν υπήρχε μια εύκολη λύση. Νομίζω ότι η προσωπική επικοινωνία όμως είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη θεσμική επικοινωνία. Τι να τα κάνουμε, τα ανακοινωθέντα τύπου και όλες τις σημαντικές συζητήσεις για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καθημερινή επικοινωνία η καθημερινή επαφή είναι αυτή που μπορεί να πείσει τους φίλους σου και τις πόλεις μας. Αυτό που κάνω και εγώ στην πατρίδα μου, στην ε, πόλη μου, στη γειτονιά μου. Αυτό είναι. Και όλα αυτά τα μικρά κομμάτια του παζλ της επαφής, της προσωπικής επαφής τελικά συνθέτουν ε, μια μεγάλη εικόνα η οποία είναι πιστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που έχουμε κάνει είναι να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να βάλουν στα εθνικά προγράμματα Ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές σπουδέ και να διδάξουν, για παράδειγμα, την ευρωπαϊκή ενοποίηση ω διαδικασία στα σχολεία, να διδάξουν τι αξίε τη Ευρωπαϊκή ενοποίηση. γιατί ένα, ένας λόγος τον οποίο ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν γνωρίζουν τις βασικές αξίες, αρχές, τους θεσμούς, κανείς δεν καταλαβαίνει καν τι είναι η θέση μου, τι κάνει ένας επίτροπος. Όλοι με φωνάζουν βουλευτή ουσιαστικά. Νομίζουν ότι είμαι βουλευτή ε, που είμαι υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευση και παιδεία. Αλλά όχι, εγώ ανήκω σε ένα άλλο θεσμικό όργανο. Ποιο το καταλαβαίνει όμω τι ακριβώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο λοιπόν να διδάξουμε το θέμα του τι είναι θεσμοί, ποιε είναι οι αρχέ, οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και την ιστορία βέβαια, για την πιο μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι ότι απέτρεψε έως τώρα τον πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό το project της ειρήνης είναι το πιο σημαντικό, το πιο ωφέλιμο, η πιο σημαντική συμβολή συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή μας ζωή. And as you said, Commissioner, και όπως είπατε, Επίτροπε, το να κατανοήσουμε τι κάνει η Ευρώπη για μας είναι η μεγάλη πρόκληση να σας παρουσιάσω την Νατάλια Φιλιππόφσκα η οποία κάθεται εκεί πίσω. Να σας πλησιάσω Νατάλια. Συμμετείχατε ε, στο πρόγραμμα Discovery U Ανακαλύπτω την Ευρώπη όταν ήσασταν 18-19 χρονών. Πείτε μας καταρχάς πώς το ανακαλύψετε το πρόγραμμα αυτό. Ναι, καταρχάς να σας πω ότι θα κάτσω γιατί δεν θέλω να, να μπω στο οπτικό πεδίο κανενός. Δεν ε, είναι από έλλειψη σεβασμού. Να πω ότι συμμετείχα όταν ήμουν 19 χρονών πέρσι. Είναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται κυρίω για 18 χρονούς βέβαια. Έγινε ε, κάποια διαφήμιση στο facebook, εκεί το είδα το πρόγραμμα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιο ιό στον υπολογιστή. Γιατί πιο πολλοί Πολωνοί αυτό είπαν. Μα γιατί να μου δώσουν κάτι δωρεάν, μου χρωστάνε. Αλλά τέλο πάντων το Έκανα κλικ και ενημερώθηκα και αποφασίσαμε με την καλύτερη μου φίλη να γραφτούμε. Και πραγματικά ως τώρα είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. And thanks to discover... Και χάρη στο πρόγραμμα Ανακαλύπτω την Ευρώπη, νομίζω ότι πήγατε σε πέντε ευρωπαϊκέ πόλει. Για πείτε μα, σε ποιε πήγατε, στο Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλε και Άμστερνταμ. Εγώ μόνο στο Παρίσι είχα πει πριν, οπότε ήταν τεράστια ευκαιρία για μένα για να επισκεφτώ τη μισή Ευρώπη ουσιαστικά σε ένα ταξίδι. Και Νατάλια, για πείτε μας, αυτή η εμπειρία πώς σας έκανε να αισθανθείτε πιο Ευρωπαία. Κυρίως πραγματικά ένιωθα ότι ήμουν στο σπίτι μου. Όπου και να πήγαινα, ο κόσμος ήταν τόσο ευγενικός. Δεν ξέρω καν αν στην Πολωνία είναι τόσο ευγενικό ο κόσμο. Πραγματικά. Γνώρισα τον κόσμο, μιλήσαμε. Πραγματικά. Χρειάστηκε να δείξω και ανοιχτό πνεύμα για να μπορέσω να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους και βρήκα και άλλους ε, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Ανακαλύπτω την Ευρώπη έμαθαν τον πολιτισμό των χωρών αυτών εκ των έσω. Ενημερωθήκαμε για ευρωπαϊκά πράγματα και άλλο ξέρετε είναι να τα μαθαίνει κανείς όλα στο σχολείο, στα... στην τάξη και άλλο είναι να τα βλέπει στην πράξη και να τα ζει. Στη Γαλλία, στο Παρίσι για παράδειγμα, το πρωινό στην Πολωνία, ξέρετε, τρώμε λουκάνικα το πρωί. Είναι πολύ μεγάλο το πρωινό και πολύ παρό. Στη Γαλλία, στα εστιατόρια, παραγγείλαμε πρωινό και μας έφεραν ένα χειμώνα, καφέ, ένα κροασανάκι εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί ήταν επιτέλους κάτι διαφορετικό. Και το έζησα εγώ ίδια στο Λονδίνο τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι στην Πολωνία. Στην Πολωνία ζούμε σε αργούς νοχελικούς ρυθμούς. Στο Λονδίνο όλοι βιάζονται. Τρέχουν. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό είναι το πώς ζουν, το στυλ του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μαδρία σας αυτά και ελπίζω να κολλήσετε τον ιό των ταξιδιών και να ανακαλύψετε πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστούμε πολύ την Αταλία Φλιμπόφτκα για την ιστορία της. Uh, Αυτή είναι πρωτοβουλία το Discover You. Είναι μοναδικό διότι έχει σχεδιαστεί για νέους Εντάξει, κατάλαβα, δεν σα αρέσει πολύ να λέμε συνέχεια νέοι, αλλά μιλάμε για του 18χρονου που έχουν πρώτη ευκαιρία για να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Ναι, σχεδιάστηκε στην Επιτροπή από δύο νέου Γερμανού και την ιδέα την πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έκανε πράξη ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απευθύνεται στους 18χρονους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Πέρσι δώσαμε την ευκαιρία σε 30.000 νέους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό τζάμπα δωρεάν βάσει ενός οδικού χάρτη όπως ονομάστηκε δηλαδή με μια συγκεκριμένη ιδέα φέτος θα φτάσουμε τους 40.000 νέους και ο επόμενος γύρος θα προκηρυχθεί την επόμενη πέμπτη αν είστε 18 να το ψάξετε Ελπίζω ότι θα πετύχουμε και αυτή τη φορά. Έχουμε σταθερή χρηματοδότηση εδώ. Θα συνεχιστεί λοιπόν σίγουρα για τα επόμενα 8-10 χρόνια το πρόγραμμα αυτό. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. Ναι, ε, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Τώρα κάποιος που δεν αντέχει να μην μιλήσει, δεύτερη σειρά με την γκρι γραβέτα. Ναι, θα μιλήσω αγγλικά ε, παρόλο που θα μπορούσα να μιλήσω τη μετρική μου. Ε, Από την Ουγγαρία είμαι και μια και έχω την ευκαιρία να, μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα, να τη μιλήσω. Νομίζω ότι πιο πολλοί κόσμος εδώ θα συμφωνήσει όταν θα σας πω ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνειδητοποιούν πραγματικά ότι είναι Ευρωπαίοι και δεν μιλάω για αίσθημα του ανήκει στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις Βρυξέλλες, αλλά στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμο ότι ανήκει στην Ευρώπη. Και ότι πραγματικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ πέρα είναι νόμιμες και σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μίλησα και εγώ τη μετρική μου και απάντησα στα ουγγρικά. Και θα συνεχίσω. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολύ αντιλαμβάνονται το θέμα της Ευρώπης ως θέμα εξωτερικής πολιτικής και στην Ουγγαρία, στην ε, χώρα μας ε, οι ειδήσει ε, ασχολούνται καταρχάς με την Ουγγαρία και μετά με την Ευρώπη αλλά Πιστεύω ότι σιγά σιγά επιτελείται μία αλλαγή και όλο και πιο πολλά ευρωπαϊκά θέματα αντιμετωπίζονται ως θέματα ιστορικής πολιτικής. Στην Ουγγαρία ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το άρθρο 7 προφανώς και διάφορα συζητήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι έχουν ε, επίδραση στην ευρωπαϊκή πολιτική για την Πολωνία, για τη Ρουμανία και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια τα ευρωπαϊκά θέματα θα γίνονται αντιληπτά όλο και πιο πολύ ω ευρωπαϊκά θέματα, ως ε, θέματα εσωτερικά. Θα έχει λοιπόν ο κόσμος την αίσθηση ότι και η Ευρώπη είναι θέμα δικό τους. Indeed. Absolutely. ακριβώς. Και τώρα μια ερώτηση εκεί πίσω. Εσείς. Ναι, ναι, εσείς. Καλημέρα, είμαι Μαρκό και είμαι Γάλλος, θα μιλήσω γαλλικά εφόσον έχω τη δυνατότητα. Το 2014 ήμουν 15 και με σόκαρε η αποχή των νέων. 25% νέοι, 25% νέοι ψήφισαν. Σε κάποιες χώρες μάλιστα ήταν 8% το ποσοστό των νέων. Σε κάποιες χώρες, στην Ελλάδα, την Αυστρία, νομίζω ότι μπορεί να ψηφίσει κανείς από τα 17 ή τα 16. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν ψηφίζουμε από τα 16 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για συμμετοχή των νέων και νομίζω ότι θα ήταν ένας τρόπος για να ενταθεί η συμμετοχή εάν κατέβαινε το όριο ηλικία στα 16. Ευχαριστούμε Μαρκό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πείσουμε τις βουλές των εθνικών κρατών να ψεφίσουν ένα τέτοιο νόμο. Από την άλλη, δεν θέλω να γίνω και ο δικηγόρος του διαβόλου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η μείωση του ωρίου ηλικία θα ε, αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής νέων ε, στις εκλογές και το τι γίνεται ε, μετά με το ποιους εκλέξει. Να ρωτήσουμε όμως τους Αυστριακούς και τους Μαλτέζους, γιατί Μάλτα είναι πρώτη φορά φέτος, οπότε θα δούμε τι θα γίνει φέτος θα πρέπει να ψάξουμε αν υπάρχει συσχετισμό μεταξύ τη μείωση τη ε, ηλικία για να μπορεί να ψηφίσει κανεί και το πώ συμμετέχει κανεί στην εκλογική διαδικασία μετά και τι γίνεται με, τις, ε, με του εκλεγμένου. Ευχαριστούμε. 1-5-5. Γιατί δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Νέων. Είμαστε το μέλλον. Θα έπρεπε να μπορούμε να πούμε τι θέλουμε. Πού ξέρετε τι θέλουμε αν δεν μας ακούτε. Κάθε χώρα θα έπρεπε να έχει τους δικούς της εκπροσώπους σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Νέους. Από πού είστε, Ρουμανία. Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας ακούω. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε. Στη δική μου τη χώρα δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε αυτή την πολιτική αγωγή. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις. Δεν ξέρουμε τίποτα για την πολιτική. Ε, σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο των Νέων και οι εκπρόσωποι των Εθνικών ε, Συμβουλίων των Νέων δημιουργούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Νέων. Και όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι των νέων ε, προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Οπότε ε, κοιτάξτε τι γίνεται με τους εκπροσώπους σας στη Ρουμανία. Και μετά υπάρχει και συστηματικός διάλογος με τους ε, συνομιλητές του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τους νέους. Οπότε αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί με έλεγχο, με επικοινωνία μάλλον, ε, με του εκπροσώπου τη δική σα χώρα. Κάποιε φορέ δεν είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα, είναι σε επίπεδο κρατών μελών. Εκεί να αποταθείτε. Εσείς τους ψηφίσατε. Πρέπει να τους ε, ελέγχετε, να λογοδοτούν. Ναι, νομίζω ότι μια τέτοια εκδήλωση μπορεί να σας πείσει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ε, πολιτικής δράσης και της λήψης αποφάσεων και των νέων. Ναι, στο 33 τώρα. Ευχαριστώ. Είμαι ο Πίτερ Μέρντοβιτ από την Σλοβενία και θα ήθελα να συνεχίσω στα σλοβενικά. Εγώ συζητώ πολύ με τους άλλους νέους και έχουμε συζητήσει πολύ το ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίζει και ποιος όχι. Πολλοί λένε ότι δεν γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι κάτι πολύ απόμακρο για αυτούς. Κι όμω ε, στα προγράμματα των σχολείων θα πρέπει να προβλεφθούν ώρε διδασκαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν γίνεται κάποιο μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Γιατί να μην προβλεφθεί υποχρέωση για ε, ε, ευρωπαϊκά μαθήματα στο πρόγραμμα διδασκαλία. Λίγε ώρε. Είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν αισθανόμαστε Ευρωπαίοι και αυτό είναι ντροπή και είναι καταστροφή για όλου μα. That's what we've proposed. Αυτό προτείναμε στα κράτη-μέλη. Να προβλέψουν στοιχεία των πληροφοριών και της γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους. Αλλά τα κράτη μέλη αποφασίζουν. Παιδεία, νέοι, ε, πολιτισμός και αθλητισμός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρέμβω στα εκπαιδευτικά των κρατών μελών λόγω χάρη ή τα διευθυντικά ή το πώ θα το οργανώσουν ή τι θα περιέχει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω συστάσεις να προτείνω δράσεις στα κάτι μέλη ξέρω εγώ να διδάσκεται η ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη ή τέλο πάντων κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο μάθημα και από την άλλη, μπορώ να ξεκινήσω προγράμματα που να έχουν προσδεθέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπω το Εράσμο. Είναι ένα πρόγραμμα πολυμερού κινητικότητα. Η κατάσταση δεν είναι απελπιστική. Γιατί ας πούμε το Εράσμους, εντάξει, έχει μόνο 9-10 εκατομμύρια συμμετέχοντες ως τώρα. αλλά ουσιαστικά είναι κάτι που επιτρέπει να διδαχθούμε μέσω της εμπειρίας. Εάν τα κράτη-μέλη πάρουν όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένταξη το εράσμος θα γίνει ακόμη πιο δημοφιλές. Θα διπλασιαστεί ο προπολογισμό του. Αν είχαμε 30 δις ευρώ για 7 χρόνια θα ήταν πολύ το χρήμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε περισσότερους νέους για να ζήσουν ε, αυτή την εμπειρία ε, την εξερεύνηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στο να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης και να αισθανθούν οικία. Είναι μια ε, πολύ σταδιακή διαδικασία, αλλά όπω όλα στην πολιτική, προσπαθούμε να προχωρούμε βήμα-βήμα για να συνεργαστούν τα κάτι μέλη και σε αυτόν τον τομέα. Εσείς εκεί με τα γυαλιά. Ναι, ναι, εσείς Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Εμιλία από τη Λιθουανία. Α, με συγχωρείς. Συνέχισε, αλλά μετά υπόσχομαι στον από πίσω ότι είναι η σειρά του. Τα μπέρδεψα. Είπα, όπως είπαμε, η Εμιλία από την Λιθουανία και θέλω να μιλήσω λιθουανικά. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, manau, ką jau girdėjau daug kartų jaunų žmonių εγώ θέλω, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι άλλοι, αλλά όντω η παιδεία είναι πολύ σημαντική ε, θα πρέπει να μπει ευρωπαϊκό περιεχόμενο στα σχολεία. Αναφέρατε πως κάθε χώρα έχει ευθύνη και αρμοδιότητες για το εκπαιδευτικό της σύστημα. Ωστόσο η Λιθουανία που είναι μέλος της Ένωσης εδώ και πάνω από 10 χρόνια αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το εκπαιδευτικό ε, στις ε, περιοχές της Υπέθρου. Εγώ προέρχομαι από την πρωτεύουσα και βλέπω πως έχουμε πολλές ευκαιρίες. Ε, η πόλη μας έχει αλλάξει, προοδεύει. Όμως Ξέρω ότι ο κόσμος που ζει στις περιοχές της Υπέθρου δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες και πάλι ερχόμενοι εδώ βλέπω πως διάφορα project και δυνατότητες που υπάρχουν εδώ υπάρχουν και προσφέρονται στους νέους όμως νέοι Πιστεύω πως θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και να μπορούν να δουν τα πράγματα αυτά που γίνονται. Ναι, είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα για το μέλλον. Οι επικοδευτικέ πολιτικέ, η παιδεία, τα μικρά σχολεία, τα σχολεία στι απομακρυσμένε περιοχέ και στι περιοχέ τη υπαίθρου, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα σχολεία και η παιδεία είναι πιο ισχυρή, ο πιο ισχυρό μηχανισμό για την κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση. Εκεί όπου δεν υπάρχουν πια σχολεία, οι ευκαιρίε για κοινωνική ένταξη και κινητικότητα αποδυναμώνονται. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι από τη μια πλευρά να αυξήσουμε την χρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών ταμείων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει και βέβαια ορισμένα ειδικά project του Εράσμους και από την άλλη πλευρά έχουμε την τεχνολογική εξέλιξη, την επανάσταση της ε, πληροφορικής. Έχουμε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που λέγεται ηλεκτρονική διδημοποίηση και συνδέει τα σχολεία online. Πάνω από 600 ε, καθηγητές και πολύ περισσότεροι ε, μαθητές συνδέονται μεταξύ τους με ψηφιακές λύσεις επιγραμμικά και αυτό μπορεί να είναι μεγάλη στήριξη για τα μικρά σχολεία στις απομακρυσμένες περιοχές γιατί έχουν τη γνώση έτσι, έχουν ε, την προσωπική επαφή και είναι πολύ σημαντικό να εξασκεί κανείς ε, την γλώσσα. Και μέσω αυτών των δημοποιήσεων γίνεται αυτό. Και βέβαια σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε περισσότερα project ε, μέσα από το Εράσμους ώστε οι νέοι και οι καθηγητές που δουλεύουν ε, σε μικρά σχολεία στις περιοχές της Υπέθρου να μπορούν να ε, αναπτύξουν περισσότερο. Επίση θέλουμε τα κρατημέλη να δώσουν περισσότερη στήριξη ώστε να διατηρηθούν τα σχολεία σε αυτές τις περιοχές όπως είπατε. Ευχαριστώ. Η σειρά σας είναι τώρα το 73. Καλημέρα σας. Λέγομαι Τζέσικα. Ε, είμαι από την Πορτογαλία αλλά ζω στο Λονδίνο. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω πως το όνομα αυτής της εκδήλωσης είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ιταλία, είπε ότι δεν πρέπει να λέγεται ευρωπαϊκή εκδήλωση για τους νέους, αλλά Νομίζω πως είμαστε διαφορετική γενιά από τους παλιότερους και έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Όταν κανείς γενικεύει, ξεχνά τις ιδιαίτερες ανάγκες ε, κάποιων ομάδων. Οι ευαισθησίες. Και τώρα θα μιλήσω πορτογαλικά. Πιστεύω πως το η εισαγωγή των ευρωπαϊκών θεμάτων στα εκπαιδευτικά συστήματα και στην ύλη των σχολείων είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και η σημερινή γενιά, η νέα γενιά ε, στο θέμα της ε, ψήφου. Να μπει ας πούμε η ψήφος στα πανεπιστήμια. Αυτό θα ήταν ε, δηλαδή να εξυγχρονιστεί η ψήφος, η ευρωπαϊκή ψήφος. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται δηλαδή τι, να υπάρξουν εκλογικά κέντρα στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει αυτό να το, να το συζητήσετε με την πορτογαλική ε, κυβέρνηση. Δεν νομίζω πως υπάρχει εμπόδιο. Κάποιος είναι και απελπισμένος, πρέπει να του δώσει το λόγο. Ναι, ναι, ναι, εσείς, εσείς. Θα μιλήσω στα ισπανικά. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Χουάν, εγώ προέρχομαι από την Καντάμπρια της Ισπανίας, από το Σανταντέρ. Είναι σημαντικό ότι εμεί που ζούμε στα χωριά και στις γεωργικές περιοχές, μέσω του Εράσμους προσπαθούμε να μπούμε... Ναι. Α, δεν άκουγα, ναι, έβαλα τα ακουστικά μου, ναι, ναι, συνεχίστε. Είναι σημαντικό λοιπόν οι τοπικές κοινότητε να συμμετέχουν στα διεθνή θέματα με τους φοιτητές. Μισό λεπτό για να βάλουμε όλοι ακουστικά. Είναι σημαντικό, ξαναλέω, οι τοπικές κοινότητες ε, να μπορεί να συμμετέχουν στα διεθνή ζητήματα. Πολλές φορές δεν ενημερωνόμαστε. Εμείς θα έπρεπε και στα πανεπιστήμια μας να έχουμε ε, θέματα ευρωπαϊκά, αλλά να φτάνουν τα νέα και στις τοπικές κοινωνίες. Ε, συμμετέχουν στα θέματα όπως ας πούμε η κοινωνική ένταξη, ε, η κοινωνική ε, ολοκλήρωση. Είναι σημαντικό δηλαδή οι τοπικές κοινότητες να καταλάβουν να, να, θεωρήσουν και να καταλάβουν ότι είναι κομμάτι ο, αυτού του project. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποια είναι η σημασία του ευρωπαϊκού ε, project. Εγώ, ας πούμε, που είμαι φοιτητή, ασχολούμαι με το γεγονός ότι ε, ε, ε, επηρεάζεται η καθημερινή μου ζωή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και το τι συμβαίνει. Το Έρασμος είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα για όλα αυτά. Μπορεί έτσι να υπάρξει περισσότερη Ευρώπη στις μικρές κοινότητες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά Δυστυχώς η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη γιατί ο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο στις Βρυξέλλες, είναι ακόμα λιγότερη γιατί όταν επισκέφθηκα το Μόλεμπεκ μετά από τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις πριν από τρία χρόνια και εκεί ήρθα σε επαφή με τους εκπροσώπους ε, των κοινοτήτων των νέων του Μόλεμπεκ και εκείνοι θεωρούσαν ότι είναι πολύ, αποστα... πολύ μακρινή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το Μόλεμπεκ είναι 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο από εδώ είναι μια γειτονιά των Βρυξελών αλλά ο κόσμος εκεί θεωρεί ότι είναι εγκαταλελειμμένος και ότι είναι τελείως εκτός της Ένωσης. Αυτό λοιπόν που είναι το πιο σημαντικό σημείο, στοιχείο της αλλαγής πιστεύω ότι μπορεί να είναι ε, ο σχηματισμός μιας κρίσιμης μάζας συμμετεχόντων στο Έρασμος. Ε, όχι μόνο στο Έρασμος, σε κάθε επιτυχημένο project της Ένωσης που μπορούν αυτοί να μιλήσουν για την εμπειρία τους στον κόσμο θα μπορούσε αυτό να σημάνει μια πραγματική αλλαγή και να είναι ε, ε, μια επιτυχία της καθημερινής επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά χέρια πρέπει να διαλέξω. Το 411. συγγνωμη που χρησιμοποιώ αυτά τα νούμερα, αλλά είναι πιο εύκολο έτσι. Καλημέρα σας. Είμαι η Χριστίνα. Θα ήθελα να μιλήσω ισπανικά. Καλημέρα σα. Εγώ είμαι καθηγήτρια σε ένα σχολείο στην Ισπανία και εκπροσωπώ τα σχολεία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθα με μια μαθήτριά μου. Πολλά παιδιά είναι εδώ για να μιλήσουν. Εγώ ήθελα να ζητήσω ε, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τι δραστηριότητε μα, ώρες για να μπορέσουμε να τι υλοποιήσουμε. Άνθρωποι όπω εσεί, κύριε Επίτροπε, να έρθετε στα σχολεία να μιλήσετε από πρώτο χέρι στου ε, φοιτητέ και στου και να πείτε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σας. Έχουμε 500 εκατομμύρια πολίτες και εγώ έχω 5 χρόνια μόνο για να κάνω κάτι και για να τους, ε, τους δω όλους. Ε, δηλαδή φανταστείτε 100 εκατομμύρια το χρόνο πρέπει <laughs> να βλέπω. Ε, φανταστείτε πόσες επαφές θα πρέπει να κάνω. Συμμετέχω στο διάλογο, συμμετέχω στο διάλογο με τους νέους φοιτητές. <coughs> Μπορούμε να δώσουμε μέσα από τα κράτη-μέλη στην παιδεία. Εμείς διπλασιάζουμε τον, ε, τον ε, προϋπολογισμό του έρασμους. Για το χρόνο, ο χρόνος δεν είναι στο χέρι μου, δυστυχώς είναι πιο δύσκολο. Όμως περισσότερα χρήματα δίνονται στο Έρασμος ε, και στα project του τα επόμενα 7 ε, χρόνια ε, στον προγραμματισμό μας, δηλαδή τον οικονομικό και στα δευτεροβάθμια σχολεία θα υπάρξει κινητικότητα και περισσότερα προγράμματα κοινωνικής ένταξης και πραγματικά εκτιμώ εσάς και τις προσπάθειες των δασκάλων γιατί εσείς είστε η φάρη των μελλοντικών κοινωνιών. Σας ευχαριστώ όλους για τους δασκάλους, τους καθηγητές για τη δουλειά σας, για το έργο σας. Επίτροπε, λαμβάνω και σχόλια online. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα του ατόμου, του ανθρώπου γιατί χρησιμοποιεί ένα ψευδόνυμο Και το θέμα των υποτροφιών ε, θα πρέπει να συζητηθεί. Ναι, είναι κομμάτι του έρασμος. Ε, μέχρι τώρα το 1 τρίτο των συμμετεχόντων ε, προέρχονταν από πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα, λιγότερο εμφρονοημένα περιβάλλοντα και θα αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, θα χρησιμοποιήσουμε τον αυξημένο προπολογισμό του έρασμος ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα κοινωνικά κίνητρα, κοινωνική ευαισθησία ώστε να αυξηθεί και η κοινωνική ένταξη. Μιλήσαμε πολύ για το έρασμο. Εδώ ο Μεσαίος, είναι, ο Λούκα από την Ιταλία, είναι εδώ στην αίθουσα. του. Σε βλέπω Λούκα. Ε, γεια σου. Ο λόγο για τον οποίο είσαι εδώ στη φωτογραφία είναι γιατί εσύ συμμετείχε στο πρόγραμμα Έρασμο στο Δουβλίνο. Πρώτα απ' όλα, πε μα γιατί διάλεξε το Δουβλίνο, γιατί ξέρω ότι ήταν η πρώτη σου επιλογή. Ναι, ακριβώ, γιατί όταν ήμουν 13 συμμετείχα στο, σε ένα καλοκαιρινό σχολείο ε, στο Δουβλίνο και ερωτεύτηκα αυτή την πόλη. Όμω, στη διάρκεια των σπουδών μου Είδα ότι είχα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Δουβλίνο, στο Trinity College μάλιστα, που είναι το παλιότερο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη και έχει και μια καταπληκτική βιβλιοθήκη με μια από τις μεγαλύτερες συλλογές βιβλίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήθελα λοιπόν να πάω για να έχω την εμπειρία της ζωής στο Δουβλίνο και την εμπειρία ενός διαφορετικού πανεπιστημίου και εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά ήμουν πολύ τυχερός που βρέθηκα σε αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον. Όσοι έχουν πάει εκεί στο Trinity College και έχουν, ε, το έχουν επισκεφθεί θα ξέρουν γιατί ενθουσιάστηκε. Τι εμπειρία όμως αποκόμισες από το έρασμο μόνο σου στο Δουβλίνο. Uh, ε, σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του να συμμετέχει κανείς στο έρασμα στο Δουβλίνο είναι ότι ανακάλυψα την κοινωνία των την ένωση ας πούμε, των φοιτητών γιατί στην Ιταλία δεν έχουμε τέτοιες οργανώσεις φοιτητών έτσι μπόρεσα να συμμετέχω σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες όπως ας πούμε ε, ήμουν μέλος της ομάδας φοιτητών για την αμνηστία συμμετείχα σε ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός ε, του Πανεπιστημίου ανακάλυψα τη δημοσιογραφία Συμμετείχα στο εφημερίδα του Πανεπιστημίου ε, πήγα επίσης να βοηθήσω παιδιά να μάθουν να διαβάζουν με άλλη ομάδα. Ένα σωρό δραστηριότητε που με βοήθησαν να καταλάβω τι θέλω να κάνω στο μέλλον και ποιος θέλω να είμαι αργότερα. Η εμπειρία αυτή λοιπόν σε έκανε να αισθανθεί ε, Ευρωπαίο. Εκεί ε, καθορίστηκε η ευρωπαϊκή σου ταυτότητα. Ναι, ναι, αποφάσισα μετά το έρασμα να ακολουθήσω ευρωπαϊκέ σπουδέ. Καταρχά, γιατί είναι ίσω κάπω μπανάλο να το λέει κανεί, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο από, όλα τα μέρη τη Ευρώπη και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι πιο Ευρωπαίο, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι κομμάτι μια μεγάλη ε, οικογένεια που είναι ενωμένη και, και, και που ε, στηρίζει τι ίδιε αξίε. Είναι αλήθεια. Ε, μπορεί κανεί να νομίζει ότι είναι μόνο λόγια, αλλά είναι αλήθεια. Ε, πρέπει κανεί να το δει με τα ίδια του τα μάτια. Πραγματικά συνδέεσαι με ανθρώπου από τι διάφορε χώρε. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εμπειρία σου και για τη μαρτυρία αυτή. Δεν σταματά αυτή η ιστορία εκεί με το έρασμος. Είσαι όμως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι έχει προσφέρει το έρασμος σε τόσο πολλούς νέους στην Ευρώπη, αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ καλή μαρτυρία που δείχνει ποια είναι τα ωφέλη του έρασμους. Η, η, ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν έρχεται σε αντίφαση με την εθνική αντίθετα ε, ε, εντείνει αυτές ε, τις ταυτότητες που έχουμε ως Ευρωπαίοι και ως πολίτες των χωρών της Ευρώπης. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αξίες του έρασμος. Παρακαλώ λοιπόν να πάρετε τώρα εσείς το λόγο γιατί σηκώνετε το χέρι σας εδώ και ώρα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Αγαπητοί φίλοι μας, στην ε, έξω έχουμε πολλούς ε, νέους ε, επισκέπτες σήμερα και πραγματικά αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν και πραγματικά μπορούμε να εξηγήσουμε το τι κάνουμε. Να του δώσουμε λοιπόν ένα θερμό χειροκρότημα και σε αυτούς που είναι πίσω στα έδρανα, τους πιο νεαρούς μας φίλους. Και τώρα θα συνεχίσω στην τρική μου γλώσσα. Um, egy német amely részt Ήμουν ε, φοιτητής. μάλλον μαθητή σε ένα σχολείο στην Ουγγαρία όπου φοιτούν ε, τα μέλη της γερμανική γερμανικής κοινότητας. Και το θέμα των μειονοτήτων θεωρώ ότι είναι θέμα που μα απασχολεί ιδιαίτερω και θα έπρεπε να μα απασχολεί ιδιαίτερω. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για του νέου εκείνου που είναι από μία μειονότητα, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στι ε, χώρε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα απάντησε στα ουγγρικά. η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάντα ασχολούταν ε, ιδιαίτερα με θέματα οικονομικά ενώ με θέματα πολιτισμικά ασχολείται το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά Και υπάρχουν και πολλές συμφωνίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις εθνικές μειονότητες στα κράτη-μέλη. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ασχολούμαστε με τις μειονότητες. Έχουμε μια επιτροπή από εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι προωθούν διάφορα θέματα που αφορούν τις μειονότητες, όπως για παράδειγμα τα θέματα εκπαίδευσης. Υπάρχει και το πακέτο μειονότητας, όπως ονομάζεται. Το πακέτο μειονότητας προβλέπει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωση προτάσεων, νομοθετικών προτάσεων προς το Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για το θέμα των μηνοτήτων και νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλες ε, εξέλιξεις τα επόμενα χρόνια στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Μάλιστα, εσείς ε, με το κόκκινο στο 294. Ευχαριστώ. Σαλό το ονομάζομαι από τη Γαλλία Είμαι γαλλικά, θα μιλήσω και μιλάμε πολύ για την ευρωπαϊκή κινητικότητα και το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο είναι κάτι το πολύ ωφέλιμο για όλους τους νέους στην Ευρώπη. Εγώ μία ερώτηση έχω να κάνω. Τι γίνεται από την άλλη πλευρά της Μεσογείου με τους πρόσφυγες Μία συνάδελφος πριν από λίγο μας ε, μίλησε για το δικαίωμα ψήφου των προσφύγων. Μας είπατε ότι αυτό έχει να κάνει με τα εθνικά κράτη-μέλη. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στην απάντηση αυτή είναι το εξή. Είναι εύκολο σε εισαγωγικά να μεταθέτουμε το πρόβλημα. σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Από την άλλη, είναι, υπάρχει κάτι πολύ απλό που μπορούν να αλλάξει. Και αυτό νομίζω είναι δορμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα προγράμματα εκπαίδευσης, στα σχολικά προγράμματα, να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε χώρες με απεικιοκρατικό παρελθόν που έχουν ε, πάρει τον πλούτο των χωρών από την άλλη πλευρά της Μεσογείου και θα πρέπει λοιπόν ο ανθρωπισμός να μας οδηγήσει στις αποφάσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ερώτηση είχε να κάνει με τα δικαιώματα ψήφου και γι' αυτό λοιπόν ε, που έχω να δώσω είναι ότι αυτό είναι από τα κράτη-μέλη. Εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποιο έχει δικαίωμα ψήφου. Τα κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων και των νέων αφιχθέντων είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών και πολλά προγράμματα Erasmus Plus, ε, υποβοήθησης των ΜΚΙΟ, αλλά και των εθνικών αρχών. Ουσιαστικά αυτό έχουν ως στόχο, την κοινωνική συμπερίληψη των μεταναστών. Και στο Εράσμους επίσης να επισημάνω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα κινητικότητας ειδικό, ένα πρόγραμμα online για τις ε, χώρες Μαγκρέμπ της ε, νότιας γειτονίας. Είναι να παρέχουμε ένα ψηφιακό λοιπόν διαδικτυακό εργαλείο και έτσι από την Τενησία, το Μαρόκο, μαθητές και φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε εργαστήρια, σε μαθήματα πανεπιστημιακά online. Παίρνουν και κάποιες ε, μονάδες για τα προγράμματα αυτά. Και έτσι προσπαθούμε να αποφύγουμε όλα τα εμπόδια των θεωρήσεων που χρειάζονται και έτσι να συμμετέχουν online σε κάποια προγράμματα. Εράσμος. Υποστηρίζουμε λοιπόν κάποιες από τις χώρες της Βορείας Αφρικής ε, που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στο πρόγραμμα Erasmus Plus και θα κάνουμε πιο πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Περνάει και η ώρα, όπως τα έλεγε και ένας κάποιος κύριος Μπαρνιέ. Να κάνουμε λοιπόν τώρα πολύ σύντομες ερωτήσεις και πολύ σύντομες απαντήσεις. Είμαι η Λουτσία και έρχομαι από τη Σλοβακία. Θα τα πω σύντομα σλοβακικά λοιπόν. Έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα, πολύ ριζοσπαστικό στη χώρα μου, που έχουν ενευρηθεί και ερευνηθεί και χθε το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε να μην καταργήσει, να μην ζητήσει την ε, διάλυση του κόμματο. Για το Εράσμου, λοιπόν, και το πόσο πρέπει να συζητηθεί από του νέου ε, το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι πλέον εκτίματα αντλούν από αυτήν. ναι, είναι σοβαρό πολιτικό πρόβλημα αυτό που θέτεται. Οι νέοι προσελκύονται από ακραίες πολιτικές τάσεις. Όμως η λύση είστε εσείς. Εσείς πρέπει να τους πείσετε. Και εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να το κάνετε σε τοπικό επίπεδο πρώτα. Εσεί με το γαλάζιο σακάκι, σειρά σα. Παρακαλώ σύντομα. Και μικρόφωνο. Ναι. Είμαι ο Μαριάν Νταλμπάν από τη Ρουμανία και είμαι διδακτορικός φοιτητής. Θα μιλήσω ρουμανικά. Ναι, είναι πολύ ωραία γλώσσα, αλήθεια είναι. με τον λαϊκισμό και τον ιντιβιντουαλισμό, τον ατομικισμό. Γνωρίζουμε ότι πολλοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί σε όλες τις χώρες ας πούμε, ακόμα και στην Ιταλία, ε, ή στην Αυστρία, πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους στο θέμα των εκλογών να ψηφίσουν οι νέοι για μια ισχυρή Ευρώπη. Τη δική μας την Ευρώπη, την Ευρώπη των νέων, μια Ευρώπη όμορφη. Well, you have to tell them the... Πρέπει να τους πείτε τις ε, επιτυχημένα, τα επιτυχημένα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τι πετύχαμε, το τι έχει γίνει στη Ρουμανία λόγω χάρη, τις επενδύσεις που έχουν πέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, από το Εράσμους, από άλλα προγράμματα. Θα μπορούσε να είναι ένα συνδυασμό των πραγμάτων αυτών. Δηλαδή να πείσουμε τον κόσμο στο τοπικό επίπεδο, να ξέρουν τι γίνεται για αυτού, ποια είναι η αλλαγή στη δική του ζωή. Ε, η προσωπική επαφή κάνει την διαφορά. Ο διάλογο με του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ξέρω ότι πρέπει να μπει κανεί στη λεπτομέρεια, αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ναι, εκεί πίσω, πίσω, εσείς, εσείς, ναι. Ε, θα μιλήσω Ιταλικά. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Σήμερα η Ευρώπη δουλεύει για το θέμα των νέων και το τι δουλειά θα βρουν οι νέοι. Ε, ειδικά ε, σε εμά, στο Νότο, από τη Ρώμη και κάτω, ε, είναι πρόβλημα αυτό. Και πολύ συχνά οι νέοι καταβλύνουν το σχολείο από τα 14. Οι ευκαιρίε του λιγοστεύουν. Ακόμη και αν βάλετε μάθημα στο σχολείο για την Ευρώπη, πολλοί νέοι δεν θα φτάσουν στο το έτος που θα διδαχθεί αυτό το μάθημα αυτό. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πλησιάσουμε αυτούς τους νέους, πώς θα τους αγγίξουμε αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο, βγαίνουν εκτός συστήματος και πέφτουν θύματα της μαφίας ή αυτών που τους εκμεταλλεύονται. Πώς θα τους δώσουμε αυτόν μια ευκαιρία. Εκεί πρέπει να φτάσει η Ευρώπη, σε αυτά τα άτομα. Διότι όσοι πάνε στο σχολείο, του άλλω είναι τυχεροί. Έχουν μια κανονική ζωή. Οι, ε, τα παιδιά αυτά όμω ε, εγκαταλείπουν το σχολείο, ζουν σε συνθήκε απόλυτη φτώχεια. Πώ θα φτάσει ω αυτού η Ευρώπη. Yes, that's, that's the ναι, είναι μια πρόκληση. Γι' αυτό Το θέμα αυτό είναι στο επίκεντρο της επόμενης Ευρωπαϊκής Στατικής για τους νέους. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις ενώσεις νέων και τους εκπροσώπους των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αισθανόμαστε ότι όντω υπάρχει πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο. Πολλοί νέοι απλώς εξαφανίζονται, αγνοούνται. Δεν θέλουν να είναι μέρος της ε, κεντρικά οργανωμένης κοινωνίας. Τι να κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε τις ενώσει νέων να οργανώσουν το δικό τους τοπικό περιβάλλον ώστε να τους βρουν αυτού τους νέους. Αυτούς που απλώς ε, απομονώνονται, αλωτριώνονται, φεύγουν. Θέλουμε να τους φέρουμε πίσω στο σωστό δρόμο, να τους εντάξουμε ξανά. Ψάχνουμε λύσεις. Πάμε πίσω. Εκείνο το κοριτσάκι που την πινακίδα του. Ναι, εσείς Γεια σα, είμαι η Ναντίν. Είμαι Πορτογαλέδα, Πορτογαλίδα. Αλλά θα μιλήσω γαλλικά και πορτογαλικά. Θα ξεκινήσω από τα πορτογαλικά. Εγώ πήγα πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο και εκεί άρχισα ε, να αισθάνομαι Ευρωπαία. Εκεί ε, αρχίσαμε να συζητάμε τη σημασία των Ευρωπαίων και των πολιτών, αλλά όπω ε, ε, σωστά υπόθηκε, υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, των χωρών τη υπαίθρου και των αστικών κέντρων, αλλά και μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι οι χώρε που είναι πιο κοντά στο κέντρο, εδώ στι Βρυξέλλε, είναι πιο ευαισθητοποιημένε. Αισθάνονται πιο Ευρωπαίε από τι υπόλοιπε χώρε που είναι νοτιότερα ή ανατολικότερα στην Ευρώπη. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώ μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά και τι χώρε αυτέ τις πιο απομακρυσμένες, ιδίως σε μια τέτοια χρονική στιγμή που το ευρωπαϊκό λόγο, το ενωμένο στην ποικιλομορφία, στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται. Δίκιο έχετε, αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Διότι λόγω χάρη στη Ρωμανία, στη Βουλγαρία, Το ποσοστό υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερο υψηλό από τι άλλε χώρε που είναι πιο κοντά στο Βέλγιο. Δεν είναι απλή λύση, διότι εντάξει, αυτό που μπορούμε εμεί να κάνουμε είναι να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδε, το Erasmus, το Discovery U, το Σώμα τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε αυτό το στόχο έχουν. Να ευαισθητοποιήσουν τους νέους που είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι εγγελιοφόροι για να προβάλλουν την ευρωπαϊκή ιδέα. Νομίζω ότι βήμα-βήμα μπορούμε να πείσουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι το ευρωπαϊκό ιδεώδες δεν είναι απλώς η ενιαία αγορά ή το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά η ζωή των ανθρώπων, η ψυχή τους και η ζωή τους σε τοπική κοινότητα και σε αυτό το επίπεδο. Πω πω αισθάνομαι πολύ άσχημα γιατί βλέπω πάρα πολλά χέρια να σηκώνονται. Θα πάρουμε τρει ερωτήσει στη σειρά. Παρακαλώ τάχιστα και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπο. Εσεί, διότι περιμένετε εδώ και πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Είμαι η Άννα από το Συμβούλιο Νέων τη Ουγγαρία. Η σύντομη ερώτησή μου είναι αυτή. Πολλοί νέοι τείνουν να μιλάνε για τα προβλήματα και τι ανάγκε του, αλλά δεν παίρνουν απαντήσει και δεν βλέπουν και τι λύσει. Τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για του νέου. <clears throat> Τι λύσει μπορεί να προτείνει. Θα παίρνουν περισσότερε απαντήσει οι νέοι στα προβλήματά του. Διότι πώ θα συμμετέχουν στις εκλογέ, θα συμμετάσχουν στις εκλογές αν δεν αισθάνονται ότι η φωνή τους γίνεται ακουστή. Δίκιο έχετε. Πρέπει περισσότερο να στοχεύσουμε στην επικοινωνία. Και εξατομικευμένε απαντήσει επίσης χρειάζονται, αλλά με τα online εργαλεία μπορεί να γίνει αυτό ίσω. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Θα μιλήσω τσεχική γλώσσα. Είμαι τη Δημοκρατία της Τσεχίας. και κύριοι, είμαι Τσέχος. Και από την Δημοκρατία τη Τσεχίας αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να ξέρει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να καταλάβει την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μιλάω τσεχικά γιατί δυστυχώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή γλώσσα. Ε, δεν είμαι πολύ καλός ρήτορα, διότι όλα αυτά με συγκίνησαν πολύ και είμαι και στη έδρανο υπαριθμών 114, ε, όπως συνήθως κάθεται αγαπημένος με ευρωβουλευτής. Λέμε πώς θα ψηφίσουν οι νέοι. Ε, ε, νομίζω ότι η προσέγγιση μας είναι λάθος. Πριν πάμε με τον κόσμο στο, στην κάλπη, πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει για να μην συμβαίνουν πράγματα όπως το Brexit ακούσαμε ότι μετά το δημοψήφισμα ο κόσμο να ψάχνει στο Google τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να το έχει κάνει το κράτο, η κυβέρνηση. Αλλά εφόσον απέτυχε η κυβέρνηση, δεν έπρεπε να έχει κάπω ε, ε, ε, παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω να έχει αλλάξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μέσω των κοινωνικών δικτύων, τη πληροφορική. Να ενημερώσει τον κόσμο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εμά η ε, συμμετοχή των νέων στι εκλογέ ήταν 18% την περασμένη φορά. Το ποσοστό προσέλευση δηλαδή. Νομίζω ότι ε, θα ήταν σημαντικό ο κόσμος να πηγαίνει και σε ένα ποσοστό 50% στις κάλπες, αλλά όχι να ενημερώνεται από τους Ρώσους και ότι οι ειδήσει να λαμβάνουν από αυτές τις πηγές. Ναι, χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη μετρική σας γλώσσα στην ε, βασική σελίδα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων online. Σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα, διότι η παρουσίαση και του Ευρωκοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες χώρες, ε, οι αντιπροσωπείες μάλλον, ε, μπορούν να κάνουν περισσότερα, στην Πράγα λόγω χάρη, για να διαδίδουν περισσότερο καλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα τηλεγραφικά, τρεις ερωτήσεις για να απαντήσετε συνολικά και στις τρεις. Εσείς, 32, μην περιμένετε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ναι. Είμαι ο Κόσμο, είμαι Ιταλό, αλλά σπουδάζω και ζω στο Λονδίνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Και κάτι που με έχει επηρεάσει πολύ ω τώρα στη ζωή μου καθημερινότητα, στην καθημερινότητα είναι το Brexit. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι άποψη έχει γι' αυτό και τι θα κάνετε για να βεβαιωθείτε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που θέλουν να μετακινηθούν και να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμένουν τα ίδια. Θα είμαστε φοιτητέ όπω οι Βρετανοί. Θα έχουμε το ίδιο επίπεδο διδάκτρων και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Θα απαντηθεί το ερώτημά σα. 1-9-4. Είμαι η Λεωνία από τη Γερμανία. Θα μιλήσω γερμανικά. Μιλήσαμε για το δικαίωμα διαδήλωση, το οποίο α, χρησιμοποιούν πολλοί νέοι σε ό,τι αφορά την αλλαγή του, των ε, δικαιωμάτων για το copyright για παράδειγμα πολλοί κόσμος, πολλοί νέοι βγήκαν στους δρόμους και πολλοί απογοητεύονται ότι δεν τους ακούν αλλά πολύ απλά δεν ακούγονται οι φωνές τους δεν εισακούονται οι επιθυμίε του. Πώς μπορούμε να δώσουμε λοιπόν σε αυτού του νέου πραγματικά φωνή. Και τέλος... Και τέλος, το, εκεί στο βάθος εσείς που κοιτάτε το κινητό σας, παρακαλώ, σηκωθείτε. Είμαι Μπογκντάνα Πάσαλα και είμαι από την Βουλγαρία. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Ε, περιμένω εδώ και πολλή ώρα για να πάρω το λόγο, αλλά ξέχασα τι ήθελα να πω. Εδώ να πω ότι η χώρα μου είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι δασκάλα αγγλικών. Διδάσκω σε 18 χρόνια που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ερχοπερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές φέτος θα συμπέσουν με το απολυτήριο των νέων στην Τρίτη ηλικίου. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής. Στόχος μας ωστόσο είναι να ε, επιδιώξουμε μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης. Στη Βουλγαρία δημοκρατία πάει χέρι-χέρι με τη φτώχεια. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια. Σας απασχόλησε το θέμα των ε, εικονικών, των δοκιμαστικών εκλογών, ας πούμε. Μήπως να γινόταν κάτι τέτοιο ε, προσπάθεια και να το ζούσαν οι νέοι από την αρχή του σχολείου, ώστε όταν φτάνουν πια στην τρίτη ηλικία να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσουν. Ναι, είπαμε την ερώτηση για το Brexit, μετά το δικαίωμα διαδήλωση και μετά τις, ε, την προσωμείωση εκλογών. Ναι, για το Brexit. Δεν έχω καμιά τέλεια απάντηση, διότι αυτό θα εξαρτηθεί από τι διαπραγματεύσει. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης μετά το Brexit, του Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή, και τι θα κάνουν μετά. Δεν ξέρουμε τι σχέση θέλουν να έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιου τομεί. Υπάρχουν κάποιε ενδείξει που μα στέλνει η δική του κυβέρνηση ότι κάτι θέλουν να γίνει μας μεταξύ μα. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ τι. Δεν ξέρουμε πώ ακριβώ λοιπόν θα καταλήξει το Brexit και δεν ξέρουμε πώ ακριβώ μπορούμε να σα βοηθήσουμε και να προσπιστούμε τα συμφέροντά σα και τι προοπτικέ σα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικαίωμα διαδήλωση. Εάν κανεί δεν σα ακούει, όπω λέτε, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Η ψήφο είναι μια ενέργεια. Εάν κανεί ψηφίσει, διαμορφώνει το μέλλον. Εάν δεν ψηφίσει, είναι απόν. Δεν είναι στην κοινωνία μέλο. Από πολιτική σκοπιά. Ε, να διαδηλώσετε λοιπόν, αλλά κάποιοι υπεύθυνοι για τι αποφάσει απλώ μπορούν να παρακάμψουν την όλη φάση των διαδηλώσεων. Να πάυσουν τις φωνές των διαδηλωτών. Όμως οι εκλογές είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί κανείς να το παρακάμψει. Το δικαίωμα της ψήφου ε, είναι ε, η ευκαιρία να στηρίξει κανείς ένα σκοπό στον οποίο πιστεύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμμετάσχει κανείς. Τώρα, σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα υπάρχουν μαθήματα για το Σύνταγμα ή για τη συνταγματική τάξη ή για τα πολιτικά δικαιώματα, η την αγωγή του πολίτη. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα υποστηρίζω όλες αυτές τις προσπάθειες που αναφέρατε. Να προβλεφθεί αυτό το μάθημα γνώσης και εξοικείωσης με το πολιτικό σύστημα, διότι η δημοκρατία χρειάζεται ενημερωμένους και ευσυνείδητους υπεύθυνου και αυτάρκης αυτών ανεξάρτητους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Μια τελευταία ερώτηση. Την πήρα από το Twitter. Ένας από τους σκάουτς που μας παρακολουθούν ρωτάει τι ελπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ερχόμενη πενταετία. Το όραμά σας για το μέλλον. Τι ελπίζετε εσείς δηλαδή ο ίδιο για το μέλλον. Ε, ελπίζω ότι θα βρούμε μια καλύτερη ε, λύση για το μέλλον της Ευρώπης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελέσματα για το ζωή των πολιτών. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες ως Ευρωπαίοι. Όλες τις ευκαιρίες που διαθέτετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Με συγχωρείτε όσοι δεν μπορέσατε να λάβετε το λόγο. Ήταν φανταστικό που είχαμε τέτοια συμμετοχή και τόσο ενεργή συμμετοχή. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους ε, ερωτώντες, ευχαριστώ τον Επίτροπο που βρήκε το χρόνο για να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε για αυτό το διάλογο. I think the conclusion is that we need... Νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να γίνονται πιο συχνά τέτοιοι διάλογοι, γιατί αποκαλύπτουν πολλά πράγματα. Παρακαλώ να μην φύγετε από την αίθουσα ακόμα, γιατί θα κάνουμε μια ομαδική φωτογραφία ως ενθύμιο ε, μιας, ε, μιας ε, ε, ιδιαίτερης μέρας έχω κάποιες ε, οδηγίες από το φωτογράφο όσοι κάθεστε άκρη-άκρη λοιπόν να συγκεντρωθείτε προς το κέντρο να γεμίσουμε όλες τις θέσεις ακόμα και τις κενές και να σταθείτε και όρθιοι στους διαδρόμους δεν πειράζει τι θέλουμε εδώ στο κέντρο είπατε παρακαλώ λοιπόν συμπτυχθείτε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 Yeah. <laughs> Are you happy? Thank you everyone and see Ωραία λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Θα τα πούμε αργότερα και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις.